Colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε μετά από αυτή την εντατική εβδομάδα ακροάσεων, μηνιακροάσεων, ψηφοφοριών. Ας επανέλθουμε στις συνήθειες εργασίες μας. να θεωρήσουμε εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Αποφάσεις από την τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών. Σημείο 1. Οι συντονιστές συμφώνησαν με την πρόταση να έχουμε άτυπη ακρόαση με τους υποψηφίους για την θέση της Προεδρίας του ΕΦΡΑΚ. και επίσημη ψηφοφορία, επίσημη ακρόαση με την Επιτροπή που θα ψηφίσει. Επίσης, ε, λαμβάνεται υπόψη το αίτημα της Άλντε να σεβαστούμε την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων και να επαναλάβω το αίτημα μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει ένας κατάλογος με υποψηφίου, shortlist και όχι ένα και μόνο όνομα που να προταθεί για την έκθεση ιδιαίτερης πρωτοβουλίας για, το, για, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά, για τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς θα προχωρήσουμε αμελητή με τον τίτλο Έκθεση Ιδίας Πρωτοβουλίας για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών και ρυθμιστικών ιδρυμάτων και φορέων. Τρίτον, οι συντονιστές ζητούν από τη Γραμματεία να προετοιμάσει και να αποστείλει κατεπίγουσα επιστολή στον υποψήφιο πρόεδρο Γιούνκερ που να του ζητήσει διευκρινήσεις για τη σχέση μεταξύ αντεπροέδρων και επιτρόπων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και επίτα οι συντονιστές ζητούν κατά τη δικασία αξιολόγησης να αποστείλουμε και μια δεύτερη επιστολή βάσει των απαντήσεων του Πρόεδρου Γιούνκερ επί του θέματος. Έπειτα, ηλεκτρονική επιτροπή και ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, η committee και οι meetings, νέα εργαλεία που είναι μέρος του ε, συστήματος ε, άνευ χάρτου για την μείωση κατανάλωσης ε, χάρτου και εγγράφων από το προσωπικό μας και τους συναδέλφους και την διεξαγωγή των συνεδριάσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Το e-committee ε, παρέχεται στο εσωτερικό διαδίκτυο και υπάρχει πρόσβαση για όλες τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές και βάσει των κατεξουσιοδότηση πράξεων και εφαρμοστικών μέτρων για τις εργασίες της Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων. Όλες οι πληροφορίες για τα ειδικά αυτά μέτρα είναι διαθέσιμες περιλαμβάνει μόνο ημερήσει διατάξεις και ε, έγγραφα το εργαλείο αυτό και θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση στα μέλη της Επιτροπής μας στο προσεχές μέλλον. Έπειτα, να σα ενημερώσω ότι ξεκίνησαν δραστηριότητες τριμερών διαλόγων. Ο πρώτος τριμερή ο τριμερής διάλογος για την ε, καταπολέμηση των ταχύων μεταφορών την 5η στι 9 Οκτωβρίου για τις ταχείες μεταφορές και την, ε, ε, λεύκανση, την καταπολέμηση λεύκανσης παρανόμων προσόδων με τη διαδικασία fast track και κάποιες ειδικές διατάξεις για την οδηγία καταπολέμησης της λεύκανσης. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με την ε, διεθνή με μια σειρά από ειδικά μέτρα. Ο επόμενο τριμερή διάλογο θα λάβει χώρα την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου το απόγευμα, 3 με 6.30 το απόγευμα. Αύριο θα ξεκινήσουν οι εργασίε μα για το ΕΛΤΙΒ, το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων. Εισηγητή για το ΕΛΚ ο κ. Λαμασούρ, ο κύριος... Κόφορτ για, το, ε, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Καμάλ, ο κύριος Ρούμπι Ροντρίγκες Βάστιες, ο κύριος Λάμπερτ, από την ΕΦΤ ΕΕ δεν έχουμε ακόμη όνομα, 14 Οκτωβρίου, 5 Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου επόμενες συζητήσεις. Και τέλος, η ομάδα εργασίας για την Τραπεζική Ένωση. Οι συντονιστές συμφώνησαν ότι η ομάδα εργασίας για την Τραπεζική Ένωση θα αναλάβει ευθύνες για την, και για την ομάδα SSM θα περιλαμβάνει 50 μέλη, 15 μάλλον μέλη βάσει του κανόνα DEONT 15 μέλη στην ομάδα εργασία. Θα τα βρείτε αυτά και γραπτός. Οι συντονιστές ενέκριναν τις διατάξεις για την έγκριση των κατεξοδότηση ε, πράξεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ε, διατεθεί στα μέλη και διατίθενται και στο ε, e-committee. Στην βάση δεδομένων για το e-committee. Ωραία. Τώρα να εγκρίνουμε το σχέδιο χρονοδιαγράμματος για το 2015. Σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης. Θα βρείτε στους φακέλους σας το σχέδιο. Να θεωρήσουμε ότι το εγκρίνεται. Ωραία, ευχαριστώ. Και τώρα να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση και συζήτηση για την επανεξέταση για την συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εισηγητής είμαι εγώ ίδιος, ο πρόεδρος. Να ξεκινήσω ευθύ αμέσω την παρουσίαση. Καλωσορίζω τις συστάσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που προτείνω την αναθεώρηση του κανονισμού 2533 του 1998 με στόχο να καλυφθούν οι νέε εποπτικέ αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως όλοι γνωρίζετε, αυτό αφορά την προληπτική εποπτεία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τι πολιτικέ του. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έχει πλήρε εποπτικέ αρμοδιότητε βάσει του κανονισμού τη 4 η Νοεμβρίου τη φετινής χρονιά. Για να, για να καλυφθούν αυτέ οι νέε αρμοδιότητε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρότεινε κάποιε. Ε, διορθώσεις στον κανονισμό του 1998 σε τρία βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζας να χρησιμοποιεί εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες για τις επιδόσεις των νέων εποπτικών, προληπτικών εποπτικών της λειτουργιών και ο στόχος είναι να μειωθεί το συνολικό άρθρο και να ε, συλλέγονται μόνο μία φορά τα απαραίτητα δεδομένα. Δεύτερον, η άδεια για την μετάδοση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών για την ε, εξάσκηση των προληπτικών εποπτικών λειτουργιών είναι κάτι που ανατίθεται πλέον στα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και τρίτον, το, η άδεια για την αποστολή των εμπιστευτικών αυτών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τις αρχές και τους φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνοι για την ε, εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού ε, Μηχανισμού Σταθερότητας. Ως εισηγητής, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας διαβούλευσης, Αυτό λοιπόν που προτείνουμε είναι να δώσουμε αυτό το δικαίωμα στην ε, αποστολή των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που είναι απαραίτητο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών αλλά μόνο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Διότι μόνο η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει αυτές τις αρμοδιότητες και όχι όλο το σύστημα. Έπειτα είναι καθοριστική σημασία να εξισορροπήσουμε την αποστολή εμπιστευτικών δεδομένων στις ε, αρχές τις υπεύθυνες αρχές, εφόσον αυτές έχουν την άδεια να λάβουν όλες τις τεχνικές και διοικητικές προβλέψεις, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη προστασία των ε, εμπιστευτικών αυτών πληροφοριών. Αυτού του είδους η απέτηση ήδη έχει προβλεφθεί από το 2009 για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και για την αποστολή των εμπιστευτικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Αυτό που ζητούμε δηλαδή είναι ήδη στον κανονισμό να υπάρξει ένας γενικός ορισμός για τις απαιτήσει του πώς εξετάζονται αυτά τα εμπιστευτικά, αυτά τα εμπιστευτικά δεδομένα και κάτι ακόμη που θα ήθελα για το οποίο θα ήθελα να τοποθετηθούν τα μέλη είναι το να συμπεριληφθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ESM Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται αυτή η συμπερίληψη. Μπορεί να έχει νόημα για λόγους backstop, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε και ακόμη και ως εισηγητής δεν το ε, κάλυψα αυτό οριστικά. Θέλω, θα ήθελα και τη δική σας γνώμη και επίσης να πω στα μέλη της Επιτροπής ότι πριν λίγα λεπτά έλαβα την αγνοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά την τοποθέτηση βλέπουμε να πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση με τη δική μας την ε, αξιολόγηση του θέματος για την ενδυνάμωση των απαιτήσεων προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποβάλλει συγκεκριμένες τροπολογίες στο κείμενο. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις διευκρινίζει περισσότερο κάποια ζητήματα από ό,τι και εγώ ίδιος ως εισηγητής για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. Αυτό λοιπόν θα θέλαμε να το συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ σκοπεύει να προβλέψει αυστηρότερε απαιτήσει. Αυτέ είναι οι γενικέ γραμμέ τη έκθεση. Και τώρα να δώσω το λόγο στου κοιόδη εισηγητέ. Ο κύριο Μπάλτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Πρέπει να σας πω που στηρίζω τις, ε, την πρόταση αυτή, ε, ολόκληρη την πρόταση έτσι όπως την έχετε περιγράψει εσείς ε, κύριε Πρόεδρε, που είστε ταυτόχρονα και εισηγητής και τουλάχιστον στο σκέλος που αφορά στον απόρριτο χαρακτήρα των δεδομένων. Παρ' όλα αυτά, ανησυχώ για κάποια θέματα στα οποία θέλω να σταθούμε μερικά λεπτά γιατί ενδεχομένως τελικά ο όγκος των πληροφοριών να είναι μεγάλος, άρα λογικό θα ήταν να ασκήσουμε κάποιο είδους αναλογικότητα. Αυτό συμβαίνει και με άλλα νομοθετικά μέτρα, τα οποία ψηφίζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια και νομίζω ότι εδώ σχετίζεται ε, το θέμα σας ε, με την αναλογικότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως όσοι έχουν την υποχρέωση αυτή υποβολής εκθέσεων ή ε, αναφοράς να μην επιβαρύνονται υπερβολικά από όλες αυτές τις απαιτήσει. Γιατί αν χρειάζεται να υποβάλεις αναφορές μέσω διαφορετικών οδών και σε διαφορετικούς φορείς και αρχές, ε, τότε καταλήγεις σε ε, επικαλύψεις, κάτι το οποίο έχουμε αποφύγει στις τομιακές οδηγίες. Και νομίζω ότι μέσω αυτής της τραπεζικής νομοθεσίας δεν θα πρέπει από κάποιο παραθυράκι να εισάγουμε αυτή την υπερβολική υποχρέωση αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω λοιπόν την ευκαιρία ε, στην αντιπροεδρία μας ε, που ε, εκπροσωπεί την ECR και που πλέον είναι και υπουργό στην κυβέρνηση του Βελγίου. Οπότε έχουμε και υπουργό οικονομικών εδώ, είχαμε και υπουργό εξωτερικών ε, Υπουργού Εξωτερικών και Οικονομικών Μάλτας και Ισπανίας. Έχουμε ανάμεσά μας και έναν επίτροπο από την Επιτροπή μας, οπότε θα ήθελα να συγχαρώ ε, τον συνάδελφο από το Βέλγιο, ο οποίος θα αντικατασταθεί από την ΚΕΙ. Ναι, και βεβαίως ε, σα ευχαριστώ πολύ. Δεν θα τα καταφέρω τόσο καλά ως ο συνάδελφο από το Βέλγιο, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον για την ε, σχετική έκθεση συμφωνούμε απόλυτα με τα όσα έχει προτείνει ο συγητής. Οπότε εδώ τουλάχιστον δεν έχω κανένα πρόβλημα. Χρειαζόμαστε κάποιο τυποποιημένο φορμάτ. Αυτό θα διευκολύνει τι μικρότερε επιχειρήσει που πρέπει να περάσουν από όλα αυτά τα κανάλια και νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει τη ροή πληροφορία ε, μεταξύ του ενιαίου επιπτικού μηχανισμού ε, που ε, εφαρμόζει όλα αυτά και τους υπόλοιπους ρυθμιστές που υπάρχουν στο σύστημα. Οπότε πρόκειται για ένα απαραίτητο βήμα που θα διευκολύνει όλους. Στηρίζουμε απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κόρα Νιούβαν Χάουζεν από ε, του φιλελεύθερου είναι η επόμενη μελήτρια και εμεί στηρίζουμε την πρόταση αυτή. Έχω απλώ μία μικρή ερώτηση για τη δεύτερη τροπολογία που υποβάλλεται και αυτό προ διευκρίνηση. Δηλαδή, σε μία από τι τελευταίε προτάσει γράφει το εξή. Έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανικά οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη φυσική και λογιστική προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Τι ακριβώ εννοείται. Αυτή η λογική προστασία. Σε τι ακριβώς αναφέρεται. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος θα απαντήσω τις ερωτήσεις. Επόμενος ομιλητής είναι η Μαρίζα Ματίας από την ΚΟΕ. is not here. Δεν είναι η κυρία Λείπει η κυρία Ματίας, δεν ξέρω αν η ΚΟΕ έχει ορίσει κάποιον άλλον να λάβει το λόγο για να σχολιάσει την έκθεση. Δεν βλέπω κάποιον, να περάσουμε στους πράσινους. Δεν είναι στην αίθουσα ο συνάδελφος, οπότε και οι πράσινοι δεν θα μιλήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Η FDD, έχετε κάποιον Δεν νομίζουμε ότι θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό αυτή η πρόταση, οπότε δεν έχουμε να σχολιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν έχουμε Άλλου συναδέλφους να ζητούν το λόγο. Μπορούμε να κλείσουμε στο σημείο αυτό, ευχαριστώντας τους ε, σκιώδεις για τις πολύ σημαντικές τους παρατηρήσεις και την δική του συνεισφορά. Μιλήσαμε για την ε, επικουρικότητα ή την αναλογικότητα αν θέλετε. Το είπε ο συνάδελφος, θα το κοιτάξουμε. Ακούσαμε και κάποιο θέμα από τους φιλελεύθερους ο ορισμός προκύπτει από το άρθρο 8α του κανονισμού που τροποποιούμε. Άρα λοιπόν πρόκειται για έναν ε, συνηθισμένο στάνταρτ ορισμό, τον οποίο απλώς αντιγράφουμε έτσι ώστε να έχουμε τα ίδια εχέγγυα ε, που εξασφαλίζονται και στα υπόλοιπα τμήματα του κανονισμού αυτού. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε στο σημείο αυτό. Έχουμε τις καταληκτικές προθεσμίες 17 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι για τις τροπολογίες. Θα τα συζητήσουμε αυτά είτε στις 3 είτε στις 4 Νοεμβρίου. 11 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε. Και βεβαίως θα περάσει και από την Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Να περάσουμε στο σημείο 5 της μερίσας διάταξης. Είναι η δεύτερη έκθεση διαβούλευσης για θέματα της ΕΚΤ που είναι η επιβολή κυρώσεων. Η εισηγητή εδώ είναι και πάλι ο νέο Υπουργό Οικονομικών των Βελγίου. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την ομάδα ECR, εάν έχουν αντικαταστήσει το συνάδελφο, φαντάζομαι είστε εσεί και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ να με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, γιατί το φάκελο αυτό δεν το γνωρίζω τόσο καλά όσο ο πραγματικός εισηγητής, οπότε Ίσως την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε τις τροπολογίες να είμαι πιο άνετη. Αυτό που θα σας παρουσιάσω εδώ είναι τα ευρήματα και η έκθεση όπως προέκυψαν από τον τότε εισηγητή, τον κύριο Φαν Overtveld, που είναι στο Eurogroup αυτή τη στιγμή, ο οποίος λοιπόν θα συζητάει τα θέματα αυτά, αλλά έχοντας διαφορετική αρμοδιότητα. Είναι σίγουρα πολύ έτοιμος για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει. Ξέρω πως κάθεται από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, αλλά είμαι σίγουρη πως θα το καταφέρει. Λοιπόν, ε, από την στιγμή που πέρασε ένας χρόνος από την πρόταση για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, ε, πρέπει να σας πω πως από την από το Νοέμβριο και μετά θα είναι σε πλήρη εφαρμογή. Και εδώ διευρύνουμε τις αρμοδιότητες που υπάρχει να επιβάλλει ο μηχανισμός αυτός ε, κυρώσεις. Ε, σύμφωνα βέβαια και με τα όσα έχουμε στον κανονισμό του Συμβουλίου. Με τις τροπολογίες που προτείνονται συμφωνεί ο εισηγητής, αλλά υπάρχουν εδώ κάποιες προσθήκες του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε το κανονιστικό πλαίσιο να είναι πιο συνεκτικό και συνεπές. Ε, έχουμε εδώ τρεις τροπολογίες που προτείνει ο κύριος Βαν Overheld. Πρώτα απ' όλα, πλαίσια του κανονισμού ε, ε, αυτού και ε, κατόπιν των εκκλήσεων, των συνεχών εκκλήσεων του Κοινοβουλίου Ζητά ο εισηγητή η απόφαση λήψη αποφάσεων να γίνεται με πιο διάφανο τρόπο. Δηλαδή, θα πρέπει ο γενικό κανόνα να είναι πω οι αποφάσει που, θα που θα επιβάλλουν ε, κάποιε κυρώσει ή πρόστιμα ε, στι επιχειρήσει να δημοσιοποιούνται. Ε, και αυτά όχι μόνο στον κλάδο που εποπτεύει, αλλά και σε περιπτώσεις που ε, ασχολείται με θέματα για τα οποία δεν έχει άμεση αρμοδιότητα υποπτική σε ε, πτώσει όπου δεν είναι ενδεδειγμένη η άμεση δημοσίευση μιας απόφασης γιατί ενδεχομένως θα ταράξει αυτή η απόφαση της χρηματοοικονομικής αγορές ή γιατί είναι δυσανάλογο αυτό με την απόφαση, τότε θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να καθυστερεί τη δημοσιοποίηση αυτών των αποφάσεων. Αλλά για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει κάποιο ρόλο και το Προεδρείο της Επιτροπής μας να ζητά να κάνει κάποιες απόρριτες ε, ε, συναντήσεις ε, για να συζητήσει πτυχές της απόφασης και βεβαίως θα πρέπει να αποδεσμεύονται οι πληροφορίες αυτές μετά από κάποιο διάστημα αυτό δηλαδή μετά από τρία χρόνια και να υπάρχει και εκ των υστέρων υποχρέωση που θα βαρύνει το μηχανισμό να εξηγήσει κάποιες αποκλίνουσες αποφάσεις. Για την μεγαλύτερη ε, διαφάνεια αλλά και για το ποιος αναλαμβάνει να κινήσει τις διαδικασίες και τις κυρώσεις επί παραβάση θέλει και εκεί μεγαλύτερη ε, σαφήνεια στην κατανομή αρμοδιοτήτων. Έχουμε το άρθρο 1α που έχουμε στις συστάσεις ε, για το μηχανισμό το χρονοδιάγραμμα για τις διοικητικές κυρώσεις. Εκεί έχει προταθεί η απόφαση να, λαμβάνει, να επιβληθεί κάποια διοικητική κύρωση ε, για μια διαδικασία παράβασης να εκπνέει πέντε χρόνια μετά ε, τη λήψη της απόφασης αυτής. Όμως, ενδεχομένως αυτό να δημιουργήσει προβλήματα σε περίπλοκες υποθέσεις, μια και καμιά φορά χρειάζεται να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκαλυφθεί μια τέτοιου είδους ε, παραβίαση. Είχε αποφασιστεί, για παράδειγμα, ε, ε, να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία όπου κινείται η διαδικασία και όχι η ημερομηνία που ε, λαμβάνει χώρα η παραβίαση των ε, κανόνων. Ο εισηγητής στη δική του έκθεση λέει πως θα πρέπει ο χρόνος παραγραφής να μειωθεί από πέντε χρόνια στα τρία χρόνια και αυτό ε, για καλύτερη διαχείριση των θεμάτων και επίσης να αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στους λόγους που θα οδηγήσουν σε αναστολή της περίοδου παραγραφής. Αυτή είναι λοιπόν η έκθεση. Την είχε ετοιμάσει ο τότε εισηγητής κύριο Βαν Overheld και πρέπει να σας πω πως τα σχόλια που θα κάνουν οι σκιώδες θα τα λάβω πάρα πολύ ε, σοβαρά υπόψη, μια και μάλλον εγώ θα χρειαστεί να αναλάβω τη γνωμοδότηση αυτή. Thank you. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε τώρα τις σκιώδες. Ο Μάρκος Φέρμπερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ που μας έφυγε ο εισηγητής μας. Τώρα από την άλλη έχει τη μοναδική ευκαιρία τα πράγματα που πρότεινε να τα εφαρμόσει ο ίδιος το Συμβούλιο. Αφού σε τελική ανάλυση πρόκειται για κανονισμό του Συμβουλίου και εμεί μόνο απλή διαβούλευση έχουμε και ακρόαση. Οπότε μπορούμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προτάσεις που δεν είναι υποχρεωμένο το Συμβούλιο να ακολουθήσει. Ήθελα να το πω αυτό εισαγωγικά και ευθύ εξ αρχή. Πολλά πράγματα είναι πολύ λογικά στην έκθεση σε ό,τι αφορά τι προθεσμίε. Δεν θέλω να μπω σε όλε τι λεπτομέρειε πλην είναι πολύ καλές ορισμένες προτάσεις. Στην πρόταση για την Κεντρική Τράπεζα να υπάρχει de facto παραγραφή όταν ανακαλυφθεί πολύ αργά μια παραβίαση. Αυτό το πρόβλημα το λύνει ο εισηγητής και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε και ελπίζω και στο Συμβούλιο τελικά να βρει αντίκτυπο. Εξ όσων ακούω από το Συμβούλιο, νομίζω πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η υπόθεση. Θέλω να σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι ως Προεδρείο της Επιτροπής ΕΚΟΝ είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ δεν ξέρω αν ε, ο εισηγητή τώρα που δεν είναι πια μέλο του Προεδρείου και είναι μέλο του Συμβουλίου αν θα μας λαμβάνει υπόψη του, συγγνώμη για αυτή την κακία, ελπίζω να υπάρξει ανταλλαγή ε, πληροφοριών και επικοινωνία. Αυτό που με ενδιαφέρει, ε, ποιος είναι αρμόδιος να επιβάλλει πλέον τις κυρώσει οι εθνικές αρχές. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβάλλονται. ποιο καλείται να τι εκτελέσει και να τι παρακολουθεί. μετά την απόφαση που λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα οι ε, Ευρωπαϊκοί οι Εθνικές Αρχές θα το χειρίζονται αυτό σωστά, ε, διοικητικά. Είναι ένα πρόβλημα. Και κάτι που με βασανίζει είναι ο κανόνας ε, για τη διαφάνεια που προτείνει ο εισηγητής. Υποθέτω ότι με τη νέα του ιδιότητα θα δείξει μεγαλύτερη συγκράτηση κάπως και θα είναι πιο επιφυλακτικός, αλλά θέλει προσοχή να μην δημοσιεύουμε πολύ νωρί αποφάσεις τη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κανονικά, όταν κάποιο υποστεί μια κύρωση, ε, θέλει να προσφεύγει εναντίον του. Οπότε να δούμε πότε θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να το δημοσιεύει αυτό η τράπεζα, να βρεθεί ε, ένας λογικός συμβιβασμός. Αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν απέχουν πάρα πολύ από τα όσα λέει ο εισηγητής, ε, ίσως βρούμε την ε, χρυσή τομή για να μην υπάρχει διπλή τιμωρία. Δηλαδή, εάν δημοσιεύονται πολύ νωρίς οι κυρώσεις, ακόμα και αν μετά από προσφυγή το δικαστήριο αποφανθεί ότι ήταν εσφαλμένη η επιβολή τους και ε, δεν έπρεπε να είχε συμβεί από την ε, πρώιμη δημοσίευση μπορεί να έχει τιμωρηθεί ήδη η χώρα από τις αγορές. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε, θα τα ε, δούμε και αργότερα και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Chairman. Και εμεί συγχαίρουμε τον εισηγητή και για την εργασία του και για το διορισμό του ε, ως Υπουργό Οικονομικό του Βελγίου. Δύο σχόλια έχουμε εμείς να κάνουμε. Ένα σημείο που ανέφερε ήδη ο συνάδελφος του ΕΛΚ έχει να κάνει με την τροπολογία 3α και κατά την άποψή μας η τροπολογία 3α δεν συνάδει με τον κανονισμό 1024 του Συμβουλίου για ιδιαίτερα το άρθρο 9 που ξεκάθαρα ορίζει για ποιος έχει τις εποπτικές και τις ερευνητικές αρμοδιότητες και εξουσίες. Όλα αυτά είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν υπάρχει εκεί χώρος για χώρις οποιασδήποτε εξουσία σε οποιοδήποτε εθνικό φορέα. Ε, το δεύτερο σχόλιο δεν είναι διαφωνία, μια ανησυχία μόνο. Και έχει να κάνει με το εξή. Παράδειγμα, η τροπολογία παριθμών 6. Αν κάποιος μπορεί Ε, να σταθεί στην απόφαση που ε, διακινδυνεύει να διαταράξει ε, την σταθερότητα των χρηματογορών. Αν υπάρχει κίνδυνος, τι λέει η εμπειρία στην πράξη. Είναι στη διακριτική ευχέρεια που μπορεί αυτό να είναι εις βάρος μικρών τραπεζών και υπέρ μεγάλων τραπεζών. Υπάρχει όρος too big to fail, ότι είναι πολύ μεγάλη μια τράπεζα για να χρεοκοπήσει. Αυτή είναι η δική μας ανησυχία σε ό,τι αφορά τα μικρά πιστοτικά ιδρύματα. Ευχαριστώ τους φιλελευθέρους. Uh, ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Άλντε θα ήθελα να διαβιβάσετε ε, ένα μήνυμα συγχαρητηρίων στον κύριο Φανόβερφελτ που ήταν αντιπρόεδρό σα και τώρα είναι νέος Υπουργό Οικονομικών του Βελγίου. Για την έκθεση αυτή καθ' αυτή συμφωνούμε με τον κύριο Φέρμπερ ότι έχει προτείνει έξυπνε λύσει ο συνάδελφο, Παραμένουν όμως κάποια ερωτηματικά για το θέμα των διοικητικών κυρώσεων Υπάρχει μια πρόταση να δημοσιεύονται στο σύνολό τους μετά από μία τριετία. Σε ό,τι αφορά και το χρονοδιάγραμμα θέλουμε πιο λεπτομερή αιτιολόγηση. Γιατί επιλέγει αυτή την τριετία, υπάρχει κανένας λόγος συγκεκριμένος, ε, μπορείτε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα και μια εκ των υστέρων υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αιτιολογεί οποιαδήποτε απόκληση. Εκ των υστέρων υποχρέωση. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, πώς και πότε θα γίνεται και με ποιο τρόπο. Και το χρονοδιάγραμμα για τις διοικητικές κυρώσεις η πενταετία λέει αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία που ελήφθη η απόφαση για διαδικασία προσφυγής ή παραβάση ε, και όχι από τη στιγμή που έχει συντελεστεί. Ο επόμενος ηγητής, η συγκήτρια προκειμένου η συγκητρια προκειμενου μπορει να μας εξηγήσει γιατί επιλέγει ε, αυτό το διάστημα. Δηλαδή όχι τη στιγμή που γίνεται ε, η παραβίαση αλλά όταν λαμβάνεται η απόφαση. Και το ίδιο ισχύει για τη μείωση της ε, περιοριστικής περίοδου από 5 σε 3 χρόνια. Αυτά, Πρόεδρε. Thank you for the e. Ευχαριστώ πολύ από την ΚΟΕ. E. Δεν έχουμε ομιλητή από τους πράσινους. Η Μαριλής. Έχω κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία ε, ευθυγραμμίζονται μετά όσα είπε η συνάδελφος αλλά ίσως έχουν άλλο στόχο. Καταρχήν για την παραγραφή. Όντως λόγω του πόσο περίπλοκο είναι οι υποθέσεις αυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε αυτά τα πέντε χρόνια, τα οποία για τον υποπτικό χρόνο δεν είναι ε, ε, αρκετά. Πιστεύω πως θα πρέπει να συνταχθεί όμως αυτή η τροπολογία με διαφορετικό τρόπο και να πούμε τα ο ένα έτος γίνεται τρία και δεν έχουμε καταληκτική προθεσμία στα πέντε χρόνια. Οπότε τελικά με τον τρόπο αυτό επεκτείνουμε, άρα το ίδιο αποτελέσμα. Στο ένα και 3, στις τροπολογίες 1 και 3 ιστορία. Μιλάμε για μια τριετή καθυστέρηση στη δημοσίευση μιας ε, κύρωσης. Όμως το 1α3 η δημοσίευση των εποπτικών κυρώσεων ακολουθεί τους κανόνες και τους νόμους της Ένωσης. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε, ε, οποιαδήποτε απόκληση από αυτούς τους κανόνες για το μηχανισμό ε, των εποπτικών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με το ένα έτος που λέμε μετά την ανείχνευση της παραβίασης και αν θα επεκταθεί αυτό στα πέντε χρόνια μετά ε, την ε, κύρωση για την παραβίαση. Ίσως θα πρέπει για κάποια ε, ευρήματα να πούμε ότι θα πρέπει ε, τα διοικητικά πρόστιμα, θα πρέπει να είναι, οι διοικητικές κυρώσεις να είναι καταναλογία με τις οικονομικές ε, κυρώσεις και βεβαίως οι κανόνες της δημοσίευσης να ακολουθήσουν το υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο. Thank you. I asked the e FTT group if... Η, η e FTT θέλει να λάβει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εμείς αναθεωρήσαμε τα έγγραφα και τα σχόλια τα οποία έχουν κατατεθεί και η δική μας ανησυχία είναι το χρονικό διάστημα το οποίο σε κάθε, σε κάθε περίπτωση επιλέγεται. Ε, αυτό που λέμε στα αγγλικά είναι ότι η δικαιοσύνη που αποδίδεται καθυστερημένα δεν είναι δικαιοσύνη. Νομίζω λοιπόν πως αν γίνει μια ακρόαση στην ΕΚΤ και μετά ε, αν αποφασίσει αυτή να επιβάλλει ε, κυρώσεις κατά κάποιας επιχείρησης, κάποιο φορέα, τι σκοπό έχει να καθυστερούμε τρία χρόνια τη δημοσιοποίηση της απόφασης ή των κυρώσεων που επιβάλλονται. Εδώ δικαιολογείται αυτό λόγω των ενδεχόμενων αναταράξεων που θα ε, προκαλέσει αυτό στις αγορές. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ε, δημιουργούμε εδώ θα οδηγήσει στο ακριβώς αντίθετο ε, αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν έχουμε συνταξιδοτικά ταμεία τα οποία έχουν επενδύσει σε τέτοιου είδους φορείς, το χειρότερο που να γίνει για ένα τέτοιο φορέο είναι να ακουστεί στην αγορά πως έχει επιβληθεί κάποια κήρυξη, αλλά κανείς δεν ξέρει ποια είναι αυτή. Μα δεν θα δημιουργήσει αυτό αναταραχή στην αγορά. Γιατί μπορεί να φαντάζει το κόσμος που η κύρωση είναι πολύ υψηλότερη από αυτή που έχει επιβληθεί. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος που δημιουργεί η μη. Ε, η δημοσιοποίηση αμέσως ε, αυτών των ε, κυρώσεων θα είναι ακριβώς οι αναταρχείς αγορές. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε, εάν έχετε σκοπό να επιβάλλετε κυρώσει και να επιβάλλετε πρόστιμα σε επιχειρήσει μέσω τη ΕΚΤ, το πιο λογικό θα ήταν να εξασφαλίσουμε πω οι πληροφορίε αυτέ δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν. Το δεύτερο που θα θέλαμε να σχολιάσουμε είναι η τροπολογία 4. Με συγχωρείτε, 3α, όπου λέει με την επιφύλαξη των υπολείπων ε, συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων των εθνικών αρμοδιών αρχών στις διοικητικές αποφάσεις κτλ. Εδώ ένα στοιχείο λοιπόν συνεχίζει και λέει μόνο σε περίπτωση που η ΕΚΤ έχει ε, του ζητήσει να κινήσουν διαδικασία για το σκοπό αυτό. Ε, δεν έχουμε εδώ πέρα όμως σύγκρουση αρμοδιοτήτων ή αποφασίζει η ΕΚΤ να ερευνήσει μια υπόθεση και μετά να επιβάλλει κυρώσεις ή είναι οι εθνικές, οι τοπικές ρυθμιστικές αρχές οι οποίες διεξάγουν την έρευνα και επιβάλλουν ε, τις κυρώσεις. Δεν μπορεί παράλληλα και οι δύο να ασχοληθούν με την υπόθεση γιατί αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση ε, και νομίζω πως το άρθρο εδώ θα πρέπει να ε, ξαναδιατυπωθεί. Η δεύτερη παρατήρηση που σχετίζεται με αυτήν είναι το τι συμβαίνει με το κατά πόσο θα πρέπει να ε, καθυστερεί ε, τα πρόστιμα η ΕΚΤ ή όχι. Ε, Εάν λοιπόν την απόφαση δεν την έχουν μάθει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οποιαδήποτε διαρροή μπορεί να χρησιμοποιήσει, να δημιουργήσει με συγχωρείτε προβλήματα στι αγορές, ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες θα παραμείνουν μυστικές και θα τις γνωρίζουν άτομα τα οποία ε, μπορούν να χειραγωγήσουν τις αγορές ακριβώς επειδή δεν δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες. Άρα λοιπόν έχουμε την οδηγία για την χειραγώγηση των αγορών η οποία εδώ παραβιάζεται. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε μία επικάλυψη από διάφορες οδηγίες που τελικά μπορεί να πλήξουν σε μεγάλο βαθμό τις χρηματογορές. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Άλλοι συνάδελφοι. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Έχουμε ακόμη χρόνο, διότι η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 5 παρατέταρτο. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, να ξαναδώσω το λόγο στην ΚΕΙ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Έχω κρατήσει λεπτομερείς σημειώσεις, το ίδιο και οι συνεργάτες μου στην αίθουσα και θα είμαι περισσότερο σε θέση να απαντήσω μόλις μελετήσω κάπω καλύτερα το όλο θέμα. Να πω πάντως ότι έχουμε δει τα διάφορα σημεία κατά και θέλουμε να δούμε κατά πόσον μπορεί να υπάρχει σύγκρουση ή όχι και κατά πόσον είναι συμβατά αυτά που προτείνονται. Μόλις τα μελετήσουμε αρκετά θα ενημερώσω και τους και εισηγητές για το αν υπάρχει πράγματι τέτοια σύγκρουση ή όχι. Συγκεκριμένα για την τροπολογία 3α. Είναι αυτό που ζητήθηκε από την ΕΚΤ και ίσως απλώς να πρέπει να αλλάξει διατύπωση για να είναι πιο σαφή τα πράγματα, για να αποφευχθεί ή οποιαδήποτε σύγκρουση. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει τροπολογία. Πάντως έχω καταγράψει όλα τα σχόλια που έγιναν και ο τρόπος που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις παραβιάσεις είναι να μην υπάρχει εκπνοή προτού αναλυφθεί δράση. Το είδα αυτό και είδα ότι ο συνάδελφος Φανόβερφελτ είχε κάνει μια πολύ καλή πρόταση αρχικά για το πώς οι κανονιστικοί περιορισμοί θα ε, μας κάνουν να αποφύγουμε να υπάρχει ακνοή της διορίας ε, πριν διαπιστωθούν οι παραβιάσεις. Πάντως είναι καθηγητής για τραπεζικές υποθέσεις και ειδικό από των θεμάτων των τραπεζών ο συνάδελφος. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, θα πρέπει λοιπόν και εγώ να ξεκινήσω καλύτερα με το θέμα. Προτού απαντήσω ε, σωστά. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ σήμερα γιατί υπάρχει και έκπιν αύριο και ομάδα εργασία σήμερα. Πάντως και το Eurogroup, οπότε θα φροντίσω να μελετήσω το θέμα για να προτείνουμε εναλλακτικέ τροπολογίε για την έκθεση και να, να προχωρήσουμε με συμβαστικέ λύσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστούμε. 17 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, λέγει προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η εξέταση τη έκθεση στι 3 ή 4 Νοεμβρίου. 11 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια, στη δεύτερη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Και πάλι να συγχαρούμε τον Γιώχαν Φανόβερφελτ για το διορισμό του και να διακόψουμε για 30 λεπτά. Συνάδελφοι, ας ξαναρχίσουμε νομίζω. Συνάδελφοι, παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Με μία δοκιμή. Άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Επτά συνάδελφοι δεν ψηφίζουν, οκτώ μάλλον. Μπορείτε να ψηφίσετε όλοι. Σχεδόν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Ωραία να ξεκινήσουμε. Θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Ντεμπάκερ, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών, εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014. Ξεκινούμε με τη συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αγκρίνεται. Συμβαστική Α1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 60. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική C Υπέρ. Κατά. Νομίζω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για έλεγχο. Άρχεται ψηφοφορία για την συμβιβαστική C. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά. Νομίζω να ψηφίσουμε για την 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο συνάδελφοι δεν ψηφίζουν. Ένας. Ένας μας λείπει. Okay, we close the vote. Πέρας της προφορίας απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Πρέπει και πάλι να ελέγξουμε για την 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. 67 υπέρ. κατά Ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 67. Πέρας. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. κατά Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 70... Η 78 λέει ο πρόεδρος ε, 74 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική D λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με δύο ψήφους διαφορά. Συμβαστική ή ε. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. 91. 91. we have 91 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία για την 91 Τέσσερις συνάδελφοι δεν ψηφίζουν. Πέρας. 9-1 πέρας. Εγώ έχω αρνητικό πρόσημο εδώ, λέει ο κύριος Φέρβερ. whip. Is adopted. Εγκρίνεται 93 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 99 άρχεται η προφορία πέρας απορρίπτεται 102 υπέρ κατά έλεγχος 102 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J. Συμβαστική J. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική K με προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Αντίρρηση, υπάρχει αντίρρηση. Πάμε απευθεία λοιπόν στη συμβαστική K, κάπα υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την K, κάπα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Και 1. Με προστίκη που προτείνει ο εισηγητής. Δεν την έχω την προστίκη. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. L2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Ωραία λοιπόν για την L2 άρχεται η ψηφοφορία. είναι σαφής η πλειοψηφία να μην κάνουμε τους ελέγχους. Ευχαριστώ. Συμβιβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική O ομικρον δύο προφορικές τροπολογίες από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες πρώτα. Αυτή να ψηφίσουμε. Κυρία Σουμπερν, με συγχωρείτε για διαδικαστικού λόγου. Ξεκινήσαμε στι 3.30 και η τροπολογία αυτή μα έφτασε στι 4 παρατέταρτο. Πώ να την έχουμε μελετήσει. Έχει ήδη ξεκινήσει η Επιτροπή μα τη συνεδριασή τη. Πώ να την έχουμε δει. Ναι, δύο αντιρρήσει λοιπόν για αυτήν την προφορική τροπολογία. Οπότε ψηφίζουμε τη δεύτερη προφορική τροπολογία από του πρασίνου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε όλη τη συμβιβαστική με, τις προφορικές, με την προφορική της τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την συμβιβαστική όπως τροποποιήθηκε προφορικός από τους πρασίνους. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά έλεγχος. Ψηφίζουμε για την 144. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T υπέρ ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα κατά τμήματα χωρίς το λόγο, τα, τους όρους The Enforcement of. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, νομίζω που να ελέγξουμε εδώ, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής T. Τα, άρχεται η ψηφοφορία, The Enforcement of, για αυτούς τους όρους. Δύο συνάδελφοι, ένας που δεν ψηφίζει, πέρα τη ψηφοφορία, απορρίπτεται. Συμβαστική U. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική W. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 100, τροπολογία 194 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική X, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική Y, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 206, 206, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Z, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.17 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ολόκληρη παραγραφός χωρίς τους όρους εν perform fatigue. Ε, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει νομίζω. Δεν μπορεί να παραμείνει έτσι αλλιώς αυτόνομο. Α, α, και α, α, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132, 231 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία 231 Πέρας. Απορρίπτεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. AC. Συμβαστική AC. Με προφορική τροπολογία από τους πρασίνους. Πρώτα θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά να ελέγξουμε για την προφορική τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική AC. Ναι, ψηφίζουμε τη συμβαστική AC χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 254. 254 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική AD υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική A, E, ΑΕ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AF υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AH υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AI, με τα ψηφοφορία που ζήτησαν οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές. Πρώτο τμήμα από το καλύπτει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος μέχρι το μείωση των εκπομπών. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, το υπόλοιπο του εδαφείου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AJ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 313, 313 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 322, 322 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Τροπολογία 332 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 338 λέει ο 338 υπέρ κατά έλεγχος 3.38 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική, αλφα όμικρον... και έχουμε μετά την προφορική τροπολογία. Θα την υπερψηφίσουμε τώρα κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ολόκληρη λοιπόν η συμβαστική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AP ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα λοιπόν στις γνώμες Εμπλό 1 υπέρ κατά. Για το εμπλό 1 θέλουμε να ανοίξουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Στις γνωμοδοτήσεις λοιπόν. Τρεις δεν ψηφίσατε. Ωραία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εμπλό 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ ξεκινάει η ψηφοφορία Δύο δεν έχουν ψηφίσει, ένας έκλεισε, εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. 6. Δεν θα ψηφίσουμε. Περνάμε στην 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 8 θα πρέπει εδώ ε, τμήματικά το πρώτο τμήμα ε, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Ξεκινάει η ψηφοφορία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4, 10, με συγχωρείτε, υπέρ. Για την 9 ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ε, νομίζω ότι έκανα εγώ λάθος εδώ το ΕΛΚ με ένα συν. Ξεκινάει λοιπόν για την 9. Έληξε. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ για το δεύτερο του 11, δεύτερο του 11 ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέσσερις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Εάν θέλετε μπορείτε να ψηφίσετε. Εάν δεν το επιθυμείτε μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Λίγοι λοιπόν. Έληξε. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Πάλι για το δεύτερο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέντε συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Έληξε. Εγκρίνεται. 14. Το δεύτερο. Το πρώτο τμήμα θα ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία λοιπόν. Εγκρίνεται. 15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 να ελέγξουμε για την 22 ηλεκτρονικά. Τρεις συνάδελφοι λοιπόν. Δύο, ένας. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Βλέπετε τα αποτελέσματα. 24 υπέρ, 23 κατά. Ήμασταν στο 22. Περνάμε τώρα στην 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται πρώτη πρόταση είναι εκτός στην 27. Η δεύτερη λοιπόν πρόταση, η δεύτερη πρόταση είναι δική του αρμοδιότητα, αλλά την πρώτη πρόταση θα ψηφίσουμε στην 27 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ανοίγει η ψηφοφορία, ξεκινάει. Λίγη. Συνέχεια ένα συνάδελφος δεν ψηφίζει, εγκρίνεται. Περνάμε στην 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά την 31. Η ψηφοφορία ξεκίνησε. Τρεις συνάδελφοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ψηφίσει. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο. 31. Υπέρ. Κατά. Μα... Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Έχουμε ήδη ψηφίσει για την 31. Περνάμε στην 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ κατά εδώ ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 45. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τμήματικά της 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά. Νομίζω ηλεκτρονικά και την 53. Ξεκινάει η ψηφοφορία. 53 λοιπόν. Λίγη. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με την ίδια. Μάλιστα, θέλετε να το κοιτάξουμε. Ωραία, ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 54. λίγη. Είχατε δίκιο. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 57, την πρώτη πρόταση. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. 57. Yes, yes. Για την υπαριθμό 57. Με συγχωρείτε. Εγώ ξεκα... λάθος. Είπα ξεκινά. Υπέρ, λοιπόν. Κατά. Ωραία. Και τότε να ξεκινήσει λοιπόν η ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Τέσσερις συνάδελφοι παρακαλώ να ψηφίσουν. Τρεις δεν έχετε ψηφίσει. Ωραία λοιπόν. Λίγοι. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο. Η 58. Υπέρ. Κατά. Και πάλι ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπάρχουν 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 63 ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία λίγη απορρίπτεται Περνάμε λοιπόν στην budget. Τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πέντε Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Την επτά Υπέρ. Παρακαλώ πολύ. Διανατάσεις χειρός υπέρ για την επτά. Άρα λοιπόν ηλεκτρονικά για την 7. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην ΙΜΚΟ, στην 20, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 ήμκο πάντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΕΝΒΙ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την ΕΝΒΙ υπαρθμών 2 ξεκινάει η ψηφοφορία Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Εγώ, λέει ο Πρόεδρος, πως έχω ως επόμενη την υπαριθμόν 4. Αλλά... So, MV4 in favor, για την 4 λοιπόν, υπαρθμόν 4, είστε υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε την MV4. Ανοίγει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέσσερις συνάδελφοι δεν ψήφισαν ακόμα. Δύο. Άρα λοιπόν κλείνουμε την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 6. Υπέρ, υπέρ της 6 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παράγραφος περιθμών 6 ένβη ξεκινάει η ψηφοφορία Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Ωραία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η εννέα υπέρ κατά ελέγχουμε την εννέα Τρεις συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει. Δύο. Ωραία. Λίγη η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Στην 10. Υπέρ. Κατά. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να καταλάβω ηλεκτρονικά για την 10. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Η 11. Υπέρ. Κατά. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 11. Έξι συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Λίγοι. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο. Η 12. Υπέρ. Και πάλι ηλεκτρονικά ξεκινά η ψηφοφορία στην 11. Ε, Στη 12 με συγχωρείτε, NV12 ξεκινά ηλεκτρονικά η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Ισοψήφισαν. Περνάμε λοιπόν στην υπαριθμό 37, το αρχικό κείμενο υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να δούμε τα εκτιμώντας. Συμβιβαστική ΑQ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. AR, ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. AS συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική AT υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. AU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32, απολογή 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική AV υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AW υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. AX υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε στη συμβιβαστική AX Τέσσερις συνάδελφοι. Τρεις, δύο, ένας. Λίγη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ισοψήφισαν λοιπόν, άρα απορρίπτεται. Περνάμε στην 37 ε, υπαριθμό τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και την τροπολογία 37. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγη. Και πάλι ισοπαλία, άρα λοιπόν απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Και πάλι ηλεκτρονικά για την 38. Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Άρα λοιπόν το εκτιμώντας αυτό δεν περνάει. Συμβιβαστική AY υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας A. Έμπλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C Εκτιμώντας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εκτιμώντας F υπέρ, κατά. Για να ελέγξουμε για το εκτιμώντας F, ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγη εγκρίνεται. Είμαστε στο H υπέρ, ε, κατά, αποχές εγκρίνεται. I υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. J υπέρ, κατά. Για να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το J, εκτιμώντας J, ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Closed. Λίγη. Is adopted. Εγκρίνεται. Περνάμε στο K, υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε λοιπόν και το K. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρα. Απορρίπτεται.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 η Αιτιολογική αναφορά 8 υπέρ, ε, το αρχικό κείμενο κατά απόχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ, κατά απόχες εγκρίνεται 15 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται η τροπολογία 6 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται η τροπολογία 7 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται έμπλ 1 η αναφορά πάντα υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ για την αιτιολογική αναφορά 1 της Ample Citation. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ήμκο τώρα, ε, το λογική αναφορά 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήμκο 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 18 κατά και 15 αποχές παρακαλώ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Exciting I would say. Συναρπαστική η ψηφοφορία πρέπει να πω. The next point. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το σημείο υπαριθμό 7. Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Θα παρακαλούσα το εξή. Όπω είδατε, είχαμε πολλέ ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε, ακόμα και για ε, αιτιολογικέ αναφορέ. Επήρε περισσότερο χρόνο από υπολογίζαμε η ψηφοφορία και τώρα θα πρέπει να επιταχύνουμε για τα αμοιβαία κεφάλαια στι χρηματαγορέ για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και το επόμενο θέμα που είναι η αιτήση έκθεση για τη φορολογία. Παρακαλώ λοιπόν να είναι σύντομοι οι και σκιώδεις. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Νίνα Γκίλ. Έχετε το λόγο. To leave the room and not to talk. Παρακαλώ, αποχωρείτε ησύχως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Γκίλ αν μπορούσαμε να έχουμε λίγη ησυχία θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Είναι η πρώτη νομοθετική πρόταση για την όλη συζήτηση που γίνεται για το παρατραπεζικό. Ε, είναι πολλοί οι διεθνείς ρυθμιστές, πολλά ε, κεφάλαια της χρήματα αγοράς, ε, ε, δημιούργησαν πολλά επεισόδια κατά τη διάρκεια της κρίσης, οπότε διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται ένα κανονικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό ήταν και θέμα των G20 και ήρθε αυτή η αντίληψη να επιβεβαιωθεί. Ε, πέρσι το Σεπτέμβριο λοιπόν ε, κίνησε αυτή η πρόταση το 2013. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ την προηγούμενη θητεία το κοίταξε αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί για διάφορους λόγους πολιτική συμφωνία και ε, το στείλε για επανεξέταση τώρα σε εμά. Θέλω να τονίσω σύντομα αυτά τα θέματα, Πρόεδρε. τι είναι τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, ποιες είναι ανησυχίες, τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς το βλέπω εγώ. Λοιπόν, πολύ σύντομα στα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς. Είναι ε, πολύ σημαντική πηγή για βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση εταιριών, τραπεζών και κυβερνήσεων. Ε, δίνουν μια ρευστότητα για βραχυπρόθεσμα για μεγάλη ε, δυνατότητα ρευστότητας, διαφοροποίησης, κεφάλαια κίνησης και τα λοιπά. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επενδυτές που τα θεωρούν ως ασφαλή ε, εναλλακτική προς τραπεζικές επενδύσεις. Να σας δώσω το πλαίσιο. Ένα τρεις ε, είναι ο κύκλος εργασιών στην Ευρώπη των αμοιβαίων κεφαλαίων, ενώ κατέχουν 40% ε, των ομολόγων βραχίας διάρκειας των τραπεζών, καθώς επίσης και των κρατών και των κυβερνήσεων. Ένα τρεις επαναλαμβάνω ευρώ διαχειρίζονται και είναι 50 συγγνώμη, 15% ε, της συνολικής χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Άρα, επιτρέπει αυτό μια ρευστότητα, ε, μια ε, κίνηση σε μετοχές για ιδιώτες, για εταιρείες, με μια μέτρια απόδοση, αλλά βράχει πρόθεσμα. Ε, και υπάρχει λοιπόν έτσι ρευστότητα, κεφάλαια κίνησης. Ε, μπορεί να είναι αντίστοιχα με τραπεζικές καταθέσεις, αλλά δεν είναι καθόλου. Ε, τι σημαίνει η ρύθμιση λοιπόν τώρα, δεδομένου των χαρακτηριστικών τους, είναι ευάλωτα στο να χάσουν επενδυτές λόγω της συστημικής τους φύσης έχουν στενή σχέση με την πραγματική οικονομία και παίζουν ρόλο στην εξασφάλιση κεφαλαίων κίνησης χρησιμοποιούν τις κεφαλαγορές ως μέσο χρηματοδότηση ε, και ε, ε, συνδέονται και με κάποιους χορηγούς που είναι μεγάλες τράπεζες, που είναι πολύ μεγάλες για να πτωχεύσουν πολύ συχνά και συχνά αυτό ενέχει ένα ενδεχόμενο ρίσκο και με ενδεχόμενη μετακύληση του κινδυνού στο φορολογούμενο. 2,1 ε, δις δολάρια έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, η σύνευ των Πολιτειών κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης. Πάνω από 200 έχουν λάβει και εξωτερική υποστήριξη για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να διατηρήσουν την αξία τους. Υπάρχει και η προστασία των επενδύσεων οι μικροεπενδυτές ε, που ε, συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες ε, πιο καθυστερημένα είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοινά πρότυπα για να είναι μεγαλύτερη ρευστότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων και να εξασφαλίζεται και η σταθερότητά τους. Πώς θα γίνει αυτό με νέους κανόνες για να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο στοιχείων ενεργητικού τόσο ημερήσιο όσο και εβδομαδιαίο για να ε, μπορεί να καταλαβαίνει ε, καλύτερα και να γνωρίζει το αμοιβαίο κεφάλαιο τον πελάτη του, το χρήστη. Με κοινούς κανόνες λοιπόν για να ε, εξασφαλίζουμε ότι τα αμοιβαία κεφάλαια ε, διαφοροποιούν ε, τη δραστηριότητά τους και επενδύουν σε στοιχεία ενεργητικού πολύ καλής ποιότητας. Για να είναι σωστή λοιπόν η ρευστότητα και σε θέση να απορροφήσει τα αιτήματα των πελατών. εμένα σαφές πλαίσιο αξιολόγησης των στοιχείων ενεργητικού όπου ε, οι εταιρείε αυτές τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν. Είναι κανονικά αμοιβαία κεφάλαια και υφίστανται τις διακοιμάσεις των τιμών. Εγώ λοιπόν τι άποψη έχω, να κοιτάξουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μια νέα αρχή για την Επιτροπή μας και υπό το φως των εξελίξεων των τελευταίων μηνών. Δύο μηνών. Στην αρχή είδαμε την ε, τροποποίηση, SEC και την ε, πρόταση της Ιταλικής Προεδρίας. Εγώ είμαι πρόθυμη να συνεργαστώ, να ακούσω, ε, συνάντησα και εξακολουθώ να συναντώ ενδιαφερομένους όταν το ζητούν. Και βεβαίως τηρώ ένα μητρό όποιον συνάντησα και όποιος θέλει είναι στη διάθεσή του για λόγους διαφάνειας. Έχω ένα κατάλογο όλων όσους συνάντησα. Ε, η αρχική μου απάντηση στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι είναι μια πολύ καλή αφιτηρία. Έχω την εντύπωση ότι τα περισσότερα άρθρα που προτείνονται δεν είναι και τόσο πολύ επίμαχα. Ε, κατά την άποψή μου, ο πολιτικός στόχος θα πρέπει να είναι ο εξής. Να αντιμετωπίσουμε το σημαστικό κίνδυνο των ε, τυχαίων ας πούμε αμοιβαίων ε, κεφαλαίων να είναι αγορά πιο ρευστή, ε, πιο σταθερή χωρίς να κινδυνεύει να στραγγαλιστεί από την υπερβολική ρύθμιση αυτός ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία για να μην ε, υπάρχει υπερσυγκέντρωση αυτής της αγοράς. Ποιο είναι όμως το πιο επίμαχο ζήτημα εδώ. Αυτό έχει να κάνει με δύο ε, είδη αμοιβαίων κεφαλαίων, ΒΙΝΑΦ και ΣΥΝΑΦ. Αυτό σημαίνει ε, ε, ότι είναι κεφάλαια που δεν ε, έχουν σταθερή αξία αλλά κειμενόμενοι με σταθερές τιμές και δίκες. Το ΣΥΝΑΦ είναι διαφορετικό Δηλαδή, όταν αγοράζει μια μετοχή ένας ε, πελάτη είναι ένα ευρώ η μετοχή, ας πούμε. Ε, ε, Παρ' όλα αυτά, μπορεί κάπως να κυμαίνεται, αλλά όχι πάρα πολύ. Δεν είναι πάντα ένα προ ένα η ονομαστική αξία. Για να αυξηθεί, λοιπόν, η σταθερότητα τέτοιου είδους αμοιβαίων κεφαλαίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες ρυθμιστικέ αρχέ και εποπτικές πιστεύουν ότι ο συστημικό κίνδυνο επιβάλλει να υπάρχει 3% ε, ένα μαξιλαράκι ε, για αποθεματικό κεφαλαίο. Ξέρω ότι θα γίνει συζήτηση εκεί για τον buffer. Αυτό είναι το πιο επίμαχο. Αυτό μου λένε όλοι. Πού θα πρέπει, αν θα πρέπει να είναι 3%. Υπάρχουν διάφορες τώρα δυνατότητες ε, και επιλογές για να το αντιμετωπίσουν. Να σας Προτείνω τέσσερις ε, τομείς και να αναλύσω. Πρώτον, να εφαρμόσουμε την πρόταση με κάποια διόρθωση ε, όπως έχει για το κεφάλαιο αυτό το αποθεματικό. Το δεύτερο είναι να αναθεωρήσουμε και να δούμε αν ένα σύστημα που βασίζεται σε ε, τέλη ρευστότητας, ρευστοποίησης, αυτό προτιμάει ο κλάδος. Το τρίτο είναι ε, να υπάρχει ένα ε, είδος ε, κειμενομένου σαν την ρύθμιση που ισχύει στις Ηνωμένε Πολιτείες για τη ρευστοποίηση. Και υπάρχει και η τέταρτη Ιταλική πρόταση που είναι ένα βίναφ με χαμηλή μεταβλητότητα. Αυτές είναι οι τέσσερις προτάσεις που εξετάζω. Αλλά η προτεραιότητα ποια είναι. Θα επανέλθω. Θα εξαρτηθεί από τις συζητήσεις που κάναμε εδώ και την ακρόαση που προτείνω να κάνουμε με τους εμπειρογνώμονες. Α, συγγνώμη, το διορθώνω. Στρογγυλή τράπεζα είναι, δεν είναι ακρόαση κανονικά. Λοιπόν, αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να ε, προσπαθήσουμε να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα για να μπορέσουν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια να βοηθήσουν σε μια καλύτερη βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Θα πρέπει να βρούμε ένα εργαλείο και μια λύση και αποτελεσματική αλλά και εφαρμόσιμη. Ε, πρέπει να πω ότι έχω κάπως απογοητευτεί μέχρι σήμερα ε, όσους έχω συναντήσει τι μου λένε. Μου λένε το πρόβλημα, κανείς δεν μου έχει πει τη λύση ακόμα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια στρογγυλή τράπεζα. Είναι χρήσιμο αυτό και σημαντικό, διότι όλοι μας θέλουμε να έχουμε μια πρόταση αποτελεσματική μπροστά μας, ε, όχι να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση. λοιπόν, τι είναι αυτή η στρογγυλή τράπεζα. Ελπίζω το σχέδιο έκθεσης 1η και 2 Δεκεμβρίου να το έχω έτοιμο. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 11η 12η. Θα συζητήσουμε στις 21 Ιανουαρίου τις ε, τροπολογίες και θα ψηφίσουμε το Φλεβάρι στην Επιτροπή και το Μάρτι στην Ολομέλεια. Δηλαδή είναι σχετικά σφιχτό το χρονοδιάγραμμα για να μελετήσουμε αυτές τις διαφορετικές δυνατότητες που έχουμε και νομίζω που ενδιαφέρονται μπορούν να συναντηθούν μαζί με μεγάλη χαρά θέλω να τους δω γιατί ε, ο κλάδος των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι σημαντικός και έχω την πρόθεση να παραμείνει και στο μέλλον. Προσπάθησα να μιλήσω όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να χωρέσω στο χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τους Γερμανείς. Και τώρα δίνω το λόγο στους σκεώδεις εισηγητές για το ΕΛΚ, ο κύριος Άγιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Καταρχάς, να συμφωνήσω με την πολύ ανοιχτόμυαλη προσέγγιση της εισηγητριάς μας, της κυρίας Ναχίλ Γκίλ, για, την, για το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό καθώς τα συνεχίζουμε την εξέταση του θέματος και επειδή έχουμε σημαντικά ζητήματα να καλύψουμε κατά τη διάρκεια τη θητεία μα, ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι να έχουν μια διαλλακτική προσέγγιση και να βρούμε συμβαστικέ λύσει για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Όχι μόνο για τον, ε, γενικότερα, για τον κλάδο αυτό, αλλά γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία, Πρόεδρε, όπω είπε και η Νίνα Γκίλ, ήδη έγινε πολλή δουλειά για το θέμα. Νομίζω ήταν πολύ λογικό που τότε δεν υπήρξε βιασύνη για να ψηφιστεί το θέμα στο Κοινοβούλιο, διότι υπήρχαν πολλά ζητήματα που έχρισαν περαιτέρω διευκρίνησης. Ο στόχος αυτή τη πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αξιέπαινο. Και το ΕΛΚ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η περαιτέρω ε, ρύθμιση των παρατραπεζικών δραστηριοτήτων Όμω, η μεταρρύθμιση των αμοιβαίων κεφαλαίων τη χρηματαγορά θα πρέπει να είναι αναλογική και να παρακολουθεί τι εξελίξει αλλού, ώστε να μην υπάρχει επιζήμια επίδραση στο πώ λειτουργούν οι χρηματαγορέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συμφωνήσω όμω, είπε λοιπόν η συγγήτρια, ότι ε, πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη προσέγγιση στο όλο θέμα. Αυτό είναι πολύ λογικό και όπω επίση το νόμα είμαστε όσο, πιο διαλεκ... όσο πιο γίνεται. Να αποφύγουμε τι επιζήμιε προτάσει που θα μπορούσε να έχει αυτή η πρόταση ως προς τη λειτουργία των αγορών. Υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία, κάποιες ε, καλοδεχόμενες ε, ρυθμίσεις που προτείνονται, όπως η διαφοροποίηση των ε, κεφαλαίων ή η επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαχείριση της ρευστότητα, οι κανόνες εποπτείας και ούτω καθεξής. Όμως με ανησυχή πρόταση να προβλεφθεί το κεφάλαιο του 3% το μαξιλεράκι του 3% που μπορεί να έχει σοβαρέ επιπτώσει για τη ρευστότητα στην Ευρώπη και να γίνει λιγότερο ελκυστική η Ευρωπαϊκή Ένωση από διεθνέ επίπεδο, από, από Μπορεί να μην είναι βιώσιμο το ανώφλη αυτό, όπω επίση για το ΣΥΝΕΦ και ΒΙΝΕΦ είναι σημαντικό αυτό και για τι χρηματαγορέ και για τα συντεκδοτικά ταμεία και για πολλέ ε, μη κερδοσκοπικέ ε, οργανώσει στι καθημερινέ του ε, δραστηριότητε. Για την φερεγγιότητα και τι αποδόσει και τη ρευστότητα, θα πρέπει το ΒΙΝΕΦ και το ΣΥΝΕΦ να χρησιμοποιούν ένα απλό επιχειρηματικό μοντέλο. τα κεφάλαια αυτά είναι σημαντικά για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τέσσερα δις χρειάζονται για το ΣΥΝΑΦ, αλλά με αυτό το όριο του 3% μπορεί να υπάρξει πρόβλημα ως προς την ε, στήριξή τους. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες μια απόφαση που απέριπτε το όριο αυτό το 3%. Και ο Επιτροπό Γκάλαγερ είπε ότι το μαξιλεράκι αυτό του 3% δεν έχει από οικονομική άποψη νόημα και ότι οι πολιτικοί ηθήνοντε θα πρέπει να ακολουθήσουν άλλη πορεία. Το 3% λοιπόν θα δίνει μια ψευδέστηση προστασία στους επενδυτές μόνον και στις αγορές και τίποτε παραπάνω. Η ιδέα του να γίνει μια κρόαση, μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπως πρότεινε η Νίνα, ε, με εκπροσώπους ε, του κλάδου και άλλους ενδιαφερομένους, είναι μια ιδέα πραγματικά ευπρόσδεκτη και θα ενθάρρυνα την Επιτροπή μας να την προωθήσει πραγματικά θα έχει νόημα να συζητήσουμε στο δυνατόν περισσότερο για την πρόταση αυτή και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της. Νομίζω επίσης χρήσιμο θα ήταν να ακούσουμε απευθείας τι θα έχει να μας πει η ίδια η Επιτροπή της Αμερικής για τις Κεφαλαγορές και να δούμε τι διαφορές μπορεί να υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών στη λειτουργία των ε, αγορών αυτών. Οι αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, λένε ότι ο κανόνας αυτός με το όριο του 3% δεν λαμβάνει υπόψη του τους περιορισμούς που έχει το διεθνές, ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο και μπορεί να δυσκολέψει τελικά τους επενδυτές. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι τα κεφάλαια ΣΥΝΑΦ μπορεί να έχουν ένα σημαντικό ρόλο για να δραματίσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία Υπάρχει η περίπτωση να είναι πολύ επιζήμια η πρόταση αυτή του 3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κεφάλαια Βίναφ και ΣΥΝΑΦ. Θα πρέπει λοιπόν, Πρόεδρε, να εργαστούμε ε, μαζί για να βρούμε ε, λειτουργικές λύσεις για το θέμα αυτό. Ευχαρίστως να συνεργαστώ με την εισηγήτρια, την κυρία Γκίλ και τους και εισηγητές τους ερχόμενους μήνες και εβδομάδες προκειμένου να βρούμε μια συμβαστική λύση για τη λειτουργία των ε, κεφαλαίων ΣΥΝΑΦ μαζί με τα κεφάλαια Βίνα. Thank you. Next speaker is the ECR Shadow Rapporteur, Mr. Και τώρα ο κύριος Καμάλα από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ, ναι, επαναλάβω αυτά που είπε ο Μπράιαν, ότι καλό θα είναι εδώ να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και διαφανείς. Διότι ήδη από την προηγούμενη θητεία το 2009 έγινε πολλή δουλειά, οπότε και εμείς πρέπει να φανούμε αντάξει. Στην προηγούμενη θητεία τα θέματα μας ε, ε, είχαν απασχολήσει έκτοτε. Για μένα λοιπόν αυτά είναι λίγο σαν να ζούμε την ίδια ιστορία ξανά και ξανά, σαν τη μέρα της Μαρμότας. Ε, διότι δεν βρέθηκαν αρχικά λύσεις για τα κεφάλαια ΣΥΝΑΦ τότε. Εδώ το πραγματικό ζήτημα είναι αυτό που ανέφερε και ο κύριος Χέις, το μαξιλαράκι για τα κεφάλαια σύνα. Ή θα λάβουμε αποφάσεις με οικονομικό νόημα είτε όχι. Το 3% λοιπόν μπορεί να κάνει το σύστημα μη βιώσιμο. Και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν θα έχει από οικονομικής άποψης νόημα ένα τέτοιο όριο. Τα περιθώρια κέρδους είναι πάρα πολύ μικρά Οπότε θα γίνουν μη βιώσιμα τα κεφάλαια με το παραμικρό όριο που μπορεί να προβλεφθεί. Θα πρέπει να δούμε και άλλες επιλογές, όπως τα όρια διάσωσης. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε με τους ειδικού όταν ε, περάσουμε στη συζήτηση της τρογγυλής τράπεζας που πρότεινε η Κινίνα. Ε, από την κρίση του 2009 είδαμε ότι τα ταμεία αυτά του ΣΥΝΑΦ πολλές φορές είχαν αντοπιστεί ως ιδιαίτερα εκτεθειμένα. Εκτίθονταν μάλιστα ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα των ε, Ηνωμένων Πολιτειών, όχι λόγω της διάθρωσής τους όμως, αλλά λόγω των επενδύσεων που γίνονται σε αυτά. Τα κεφάλαια λοιπόν ε, ΣΥΝΑΦ και ΒΙΝΑΦ δείχνουν ότι από τα δύο τα ΣΥΝΑΦ τα πάνε καλύτερα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι ασφαλή τα κεφάλαια αυτά, απλώς είναι μία λύση. Εκροέ επίση το λόγο τη κρίση υπήρξαν και στα γαλλικά βίνα και το κατέγραψε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Bundesbank ε, έπρεπε να δώσει εγγυήσεις ε, κατά τη διάρκεια τη κρίση για τα κεφάλαια αυτά. Γιατί λοιπόν ήταν τόσο εκτεθειμένα σε κινδύνου τα κεφάλαια αυτά, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα στον χρηματοδοτικό τομέα. Ε, είναι η διάρθρωσή του η ίδια ή το που επενδύονται τα κεφάλαια αυτά. Νομίζω λοιπόν σημαντικό είναι να έχουμε αυστηρέ απαιτήσει διαφοροποίηση και ρευστότητα. Αυτό συμφωνούν νομίζω και οι συγκεκριά και οι σκιώδει. Να δούμε ποια θα είναι τα όρια διάσωση και το κόστο του και την στενή ε, διασύνδεση των Αμερικανικών με τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Στην ε, αμερικανική αγορά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση προς τη λιανική. Μικροεπενδυτές να ε, ανατρέχουν στα κεφάλαια αυτά, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεσμικοί οι επενδυτές περισσότερο. Πού πηγαίνουν όμως τα κεφάλαια αυτά, θα πρέπει να πηγαίνουν απευθείας στα Βίναφ ή στον ε, συμβατικό τραπεζικό τομέα. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε είναι συστημική συγκέντρωση και υπερβολική ε, λοδιασύνδεση. Θέλουμε να υπάρχει διαφοροποίηση στον τραπεζικό τομέα και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Όχι να κάνουμε πιο ασταθή μια ασταθή κατάσταση. Και να είμαστε εδώ σαφείς. Ακόμη δεν έχουμε επιλύσει το βασικό πρόβλημα των ε, τραπεζών που ε, τελικά διασώζονται με χρήματα των φορολογουμένων επειδή αποτυγχάνουν. Εδώ πρέπει κάτι να κάνουμε και να προσέξουμε ιδιαίτερως για το εύρωστο του τραπεζικού τομέα γενικότερα. Ε, σε γενικές γραμμές συμφωνώ με την προσέγγιση της ε, εισηγήτριας, με πολλά από τα σχόλια του κυρίου Χέις και αναμένω τη συνεργασία μας για να είμαστε όσο δυνατόν διαφανέστεροι. Thank you. Now for the... Ευχαριστώ πολύ από τους φιλελεύθερους λοιπόν, ο κύριος Γέζεκ. Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια μίλησε για μια ανοιχτή προσέγγιση και πρέπει να σας πω πως και εγώ το ίδιο έκανα. Έκανα πάρα πολλές συναντήσεις με πολλούς από τους εμπλεκόμενους φορείς και πολύ συχνά διαφωνούν μεταξύ τους. Κάποιοι ζήτησαν να απαγορεύσουμε τις ε, ΣΥΝΑΒ, Υπάρχει βέβαια το θέμα με την ε, ρευστότητα, με το τίμημα ρευστοποίηση, με το μαξιλαράκι. Υπάρχουν και κάποιες φωνές οι οποίες ζήτησαν να μην κάνουμε τίποτα. Εγώ αυτή τη στιγμή σιγά σιγά βγαίνω από το δάσος και σε αυτό θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου έτσι ώστε να γίνει μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης γιατί καλό θα ήταν να ανταλλάξουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε και τα δεδομένα έτσι ώστε να καταλήξουμε. Άρα λοιπόν ανυπομονώ και εγώ να γίνει αυτή η συζήτηση και να συνεργαστούμε για τούτον εδώ το φάκελο. Από την ΚΟΕ, ποιος θε... ο κύριος Βιέγκας έχει το λόγο. Ευχαριστώ εδώ πολύ γρήγορα, μιας και βρισκόμαστε στο χώρο της αλχημίας και βρισκόμαστε στην καρδιά του προβλήματος που προξένησε την σημερινή κρίση, ε, ιδίως από το χρηματοπιστωτικό τομέα προς την πραγματική οικονομία με την ανάδυση ενός μιας αγοράς τίτλων, με προεκτάσεις που κανείς ε, δεν καταλαβαίνει και κανείς δεν καταλαβαίνει τι πουλάει και τι αγοράζει. Αυτό προφανώς μας δείχνει ότι είναι πολύ βαθιές οι ελλείψεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ότι δεν λειτουργεί και αναζητούμε επί της ουσίας πώς θα διορθώσουμε όλες αυτές, όλα αυτά τα, τις ελαττωματικές διαστάσεις της αγοράς που είναι τα βαθύτερα αίτια της κρίσης. Προφανώς είμαστε πρόθυμοι προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας στην διαχείριση της αγοράς αυτής. Ε, για την αγορά αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων. Θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη σταθερότητα και προστασία των επενδυτών. Στη συζήτηση όμως αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η ανάγκη να υπάρχει δημόσιος έλεγχος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κάτι που δεν έχει αναφερθεί αρκετά και χωρίς τον οποίο έλεγχο δεν μπορούμε και εμείς να σκεφτούμε ότι θα υπάρξει μια βιώσιμη λύση. Ευχαριστώ πολύ από τους πράσινους λοιπόν η κυρία Ζολή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω. Πρέπει, πρέπει να σας πω πως ξεκινήσαμε τη συνεργασία με την κυρία και με του υπόλοιπου γιατί θεωρούμε πω είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίσουμε τις χρηματαγορές αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουμε να συνεργαστούμε με πάρα πολλούς φορείς, όχι μόνο με το Δουνουτού, αλλά και με τα διάφορα, ε, τις διάφορες αρχές ε, στις χώρες μας, με τις ευρωπαϊκές αρχές, για να ξεπεράσουμε αυτούς τους συστημικούς κινδύνους, ε, από τους οποίους κινδυνεύει το παρατραπεζικό σύστημα. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε πως η αρχή που θα έπρεπε να μας διέπει είναι ίδιες υπηρεσίες, ίδιοι κανόνες. Ο κύριος Ελχαντράουι είχε κάνει πολλά την προηγούμενη θητεία και ελπίζω πως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε βασιζόμενοι στις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει. Για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι να έχουμε μια μεταβατική φάση έτσι ώστε να ξεκινήσουμε με τη ΣΥΝΑΒ. Με συγχωρείτε, με, έτσι ώστε να ε, κλείσουμε τη ε, ΣΥΝΑΒ γιατί ε, ξέρετε τι προβλήματα προκαλούν ε, καμιά φορά και κρίσεις πανικού που μπορεί να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την χρηματαγορά. Θα ήθελα λοιπόν να εργαστούμε με έναν τρόπο που θα μετατρέψει αυτές τις ΣΥΝΑΒ σε ΒΙΝΑΒ. Και αυτό μέσα σε μια σύντομη περίοδο, για παράδειγμα δύο χρόνια, όπως προτάθηκε φέτος το καλοκαίρι. Μια άλλη προτεραιότητα θα ήταν αυτά τα κεφάλαια να μην μπορούν άμεσα ή έμεσα να κερδίσουν ε, από το γεγονός που θα τους προσφερθεί και ένα δημόσιο δίκτυο ασφαλείας. Πιστεύουμε πως χρειάζεται βέβαια ένα ε, μαξιλαράκι που θα λειτουργεί εκτός αντίθετα με τους κύκλους της οικονομίας, γιατί αυτό θα στηρίξει. Αλλά εμείς θέλουμε να έχουμε κανόνες, για παράδειγμα, οι αμοιβέ των μάνετζερ να είναι ανάλογες με τις αμοιβέ έτσι όπως έχουν περιοριστεί στον τραπεζικό κλάδο. Τα θέλαμε λοιπόν αυτά τα ε, αμοιβαία να ξεκινήσουν με τα όσα έχει, έχουμε συμπεριλάβει στην ε, οδηγία για τα τραπεζικά και θα θέλαμε όσες από αυτές δραστηριοποιούνται σε φορολογικούς παραδείσους να μην μπορούν να θέσουν σε εμπορία τις υπηρεσίες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τον κίνδυνο ε, χρεοκοπίας και στα πλαίσια των όσων έχουμε βάλει στην οδηγία MIFID πιστεύω πως θα έπρεπε να ήταν χρήσιμο να έχουμε κάποια παράγωγα προϊόντα τα οποία είναι εγκεκριμένα προς αγορά. Κάτι τέτοιο είναι απαράτητο γιατί θέλουμε να περιορίσουμε στο μέγιστο δυνατόν την έκθεση που, έχουμε, που έχουν ε, αυτά τα αμοιβαία σε επικίνδυνα παράγωγα. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε ποιο είναι ο ρόλος που πρέπει να έχουμε, ποιο είναι ο ρόλο που θα έχει η τράπεζα και τι θα γίνει με αυτά τα αμοιβαία τα οποία έχουν γίνει σχεδόν τράπεζες. Εμείς είμαστε υπέρ του να ενισχυθεί η αρμοδιότητα που υπάρχει και να υπάρχουν μεγαλύτερες, ε, ε, περισσότεροι κανόνες που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια προς τον ε, ευρύ Και για να το κλείσω θα συμφωνήσω με τα όσα είπε η Νίνα και θα πω πως είμαι υπέρ μιας συζήτησης στρογγυλή τράπεζα. Σας ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βόλφ από την EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, τα αμοιβαία κεφάλαια αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για να ανακάμψει η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και η Νίνα, είναι τεράστια σημασία. 22% του βραχυπρόθεσμου χρέους που εκδίδουν τα κράτη-μέλη και 38% του ε, χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη. Μιλήσαμε για την νομοθεσία. Μέχρι τώρα τι είναι. Είναι πολλοί που μας δημιουργούν προβλήματα. Τα προβλήματα ε, θα αντιμετωπίσουν αυτούς που έχουν ε, την έδρα των δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, αλλά πελάτες είναι εκτός Ευρώπης. Και τελικά μήπως σηκωθούν και φύγουν. Ε, υπάρχει ένα κόστος το οποίο εμείς είναι αμεληταίο από ό,τι φαίνεται για μας και θέλουμε να συνεχίσουμε να το Διονύζουμε. Είναι κόστος και λειτουργικό και κεφαλαίο και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα ε, διατηρούν ε, στην αγορά τους φορείς. Αν κοιτάξετε το τελικό χρήση και τι επιπτώσεις θα έχει σε αυτό είναι τεράστιες. Γιατί σήμερα οι περισσότεροι που εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο είναι 2 ε, με 3% σε σχέση με τις τράπεζες οι κεφαλαίκες τους απαιτήσει ε, και αν ε, μπουν νέες κεφαλαίκες απαιτήσει ε, θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Τους ζητούμε να παρέχουν μια υπηρεσία σε πολλές εταιρείες, σε πολλές επιχειρήσεις και τώρα αν τους αφαιρέσουμε αυτό το πλεονέκτημα του κόστους θα ψάξουν καλύτερους προορισμούς. Το θέμα δεν είναι μόνο το λειτουργικό κόστος αλλά και το κεφαλαιακό κόστος που επιβάλλουμε και τι ε, θα σημάνει αυτό για το κρατικό χρέος. Θα είναι πολύ πιο ε, σημαντικό γιατί μπορεί να αποχωρήσουν συνολικά από την ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε τις ευκαιρίες δανεισμού, ιδιαίτερα ε, με τις οδηγίες που θα χειρίζεται ο Λόρδος Χιλ, είναι ανοησία να αρχίζουμε να κάνουμε αυτή την επιδρομή προς τους φορείς που δίνουν χρήματα στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να προσέξουμε τι ε, επίπτωση θα έχει ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Ε, αυτά που διαβάζω δεν με ε, κάνουν να είμαι αισιόδοξο. Είναι πολύ μεγάλες οι δυσκολίες για να βρούμε μια καλή λύση και να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι το κακό είναι ότι αυτά τα ταμεία έφεραν την κρίση. Δεν ισχύει αυτό. Ε, α, ότι είναι εικονικέ τράπεζε. Δεν είναι. Δεν έχουν λιανικού πελάτε και ακόμα και αν είχαν ε, μικροκαταθέτες. Ε, το πρόβλημα είναι στι θεσμικές τράπεζες. Ε, εκείνες δεν πρόκειται να δανείσουν περισσότερα χρήματα εάν κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Δεν θα πρέπει να σκοτώσουμε την κότα που κάνει το χρυσό αυγό στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί να τους επιβαρύνουμε περισσότερο, γιατί τους θεωρείτε εσείς ε, επικίνδυνους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τελείως διαφορετικό το μοντέλο. Εμείς αντιγράφουμε τώρα την Αμερική. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσει. Σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους τους κοιόδης για τα σχόλιά σας και πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους και Δύο πράγματα να πω μόνο για την στρογγυλή τράπεζα. Έχει σημασία να ακούσουμε την SEC, την Αμερικανική Επιτροπή Κέφαλη Αγορά. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο Brian Μπορεί να είναι δύσκολο όμως γιατί Γύρω στις 4 με 5 Νοεμβρίου το προγραμματίζουμε. Μέχρι πότε θα μπορέσουμε να τους καλέσουμε. Θα πρότεινα στη γραμματεία μια βιντεοδιάσκεψη. Όλοι οι σκιώδεις εισηγητές μαζί τους με την ε, SEC. Ελπίζω να μπορέσει να στηθεί αυτό, να οργανωθεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Και για αυτά που είπε ο Σαΐντ Καμάλ, ε, για τις εταιρείες ε, που είναι μεγαλοεπενδυτές και επενδύουν. Ποιοι είναι, πολύ θα ήθελα να τους γνωρίσω. Θα μπορούσες να με βοηθήσεις να εντοπίσω κάποιον που χρησιμοποιεί αυτά τα ε, κεφάλαια, ένα φυσικό πρόσωπο υπαρκτό να έρθει στη Στρογγυλή Τράπεζα με όλους και όδης ηγητές, για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι μεγάλοι επενδυτές που χρησιμοποιούν αυτά τα ταμεία. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Επανειλημμένα το ακούω αυτό το επιχείρημα, ότι είναι ουσιαστικό και σημαντικό για τα αμοιβαία κεφάλαια τα επενδυτικά, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ε, θα με ενδιαφέρει να συναντηθώ μαζί τους. Και άλλοι συνάδελφοι μπήκαν σε πολλές λεπτομέρειες εδώ. Ιδιαίτερα πράσινη. Με χαρά να συζητήσουμε τις ιδέες που προτείνετε αλλά όπως σας είπα, προς το παρόν αναθεωρώ και χτενίζω έτσι τις τρεις ή τέσσερις ε, εναλλακτικές ε, λύσεις που έχουμε και στην ε, ακρόαση, μάλλον μετά τη στρογγυλή τράπεζα θα συντάξω μια έκθεση προς έγκριση. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Περιμένω να συνεργαστούμε πολύ χαρά. Ευχαριστώ. Υπενθυμίζω το χρονοδιάγραμμα, Πρόεδρος συζήτηση του σχεδίου έκθεσης 1η 2 Δεκεμβρίου, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 11 11η Δεκεμβρίου, συζήτηση των τροπολογιών 21 Ιανουαρίου, ψήφιση στην ΕΚΟΝ στις 23-24 Φεβρουαρίου και ολομέλεια στη 2η του Μαρτίου. Σας ευχαριστώ και παίρνουμε στο τελευταίο θέμα που είναι η αιτήσια τελευταιο θεμα που ειναι η εκθεση για τη φορολογία και θα δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Εύα Καηλή από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ καλωσορίζω την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την ετήσια έκθεση για τη φορολογία που βεβαίως ε, μετά τις ακροάσεις περασμένης εβδομάδας αυξήθηκε σε σημασία. Ακόμα και αν οι πολιτικές ομάδες έχουν διαφορετικές θέσεις για τα θέματα της φορολογίας, είμαι πεπισμένη ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε ότι η πρόοδος θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορη, πιο αποτελεσματική και ότι θα μπορούσαμε ε, να αποδώσουμε καλύτερα και χαιρετίζουμε τα όσα είπε ο Πιχέρ Μοσκοβισή για τις ε, φορολογικές φιλοδοξίες της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια όλων των επιτρόπων είπαν ότι χρειάζεται μία ατζέντα για να μεταρρυθμιστεί το σύστημα και να είναι πιο ενσωματικό τομένο, πιο ολοκληρωμένο στην ε, οικονομική πολιτική φιλική προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μετατοπιστούμε από αυτή τη μονολυθική νομισματική πολιτική που δεν έχει καθόλου επιτύχει μέχρι σήμερα, επιτρέψτε μου να προσθέσω, προς μια πιο χαλαρή πολιτική φιλική προς τις επενδύσεις ε, και με φορολογικές ευθυγραμμίσεις και προσαρμογές. Ε, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Ε, είναι καταστροφικές και ολέθριες οι συνέπειες καθυστέρησης. Ε, δεν καταλαβαίνουμε την αντίσταση που εξακολουθεί να ισχύει ως νοοτροπία, αντιστεκόμαστε στις αλλαγές. Ελπίζω να μην είναι η πλειονότητα αυτή ποια είναι η ανάγκη για προσανατολισμό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργεί καλά και να είναι εύληπτη φορολογική πολιτική, πιο δίκαιη, πιο φιλική προς την ανάπτυξη, ε, σεβόμενη το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, σεβόμενη το δικαίωμα στην προστασία των βασικών μισθών και το δικαίωμα στο επιχειρήν. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ένα φορολογικό καθεστώς που θα μετατοπίζει ε, το βάρος της φορολογίας για να προστατεύει τους ασθενέστερους, τους μικροϊδιοκτήτες, τους εργαζομένους ε, και τη σχολάζουσα ε, περιουσία και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει αναλογικά με το πλούτο και δίκαια, με το δίκαιο που, πλούτο που παράγουν να φορολογούνται. Ο καθένας βάσει των δυνατοτήτων. Επίσης, προτεραιότητα είναι να ελέγχονται πολυεθνικές εταιρείες που φόρο διαφεύγουν. Αυτή τη στιγμή αφήνω στην άκρη τις τεχνικές λεπτομέρειες, είναι μια δεοντολογική αρχή και βάση για κοινή φορολογία που ελπίζω όλοι να συμφωνήσουμε ως ένα πρώτο βήμα. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλα θέματα που εκκρεμούν συνεχώς στις εκθέσεις μας για τη φορολογία και χρειάζεται να συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα ε, ότι δεν ε, παραγνωρίζουμε, δεν αγνοούμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροποφυγή ε, και τη φορολογική απάτη ή την επιθετική φορολογική ε, ε, πολιτική και προγραμματισμός, φορολογική παράδειση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζητήματα που καλούν σε αποτελεσματική αντιμετώπιση. Φέτος λοιπόν το έχουμε τονίσει στην έκθεσή μας και ελπίζω να είναι τελευταία φορά διότι θα πρέπει να επιτελεστεί σημαντική πρόοδο σε άλλα σημαντικά θέματα επίσης τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως είναι ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ε, η κοινή ε, ε, νομοθεσία για τη φορολογική βάση των επιχειρήσεων, εκθέσεις αναχώρα, το τραπεζικό απόρριτο και άλλα. Ε, είναι ε, απλώς ενδεικτικός ο κατάλογος των θεμάτων που σας παρέθεσα. Ε, είναι μια κληρονομιά της προηγούμενης θητείας. Θα πρέπει εμείς να δώσουμε συνέχεια και ήρθαμε να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα και άλλα και παραγωγικά και ρεαλιστικά για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τους συναδέλφους για τα θέματα που θεωρούν πιο σημαντικά ώστε να συμπεριληφθούν στην έκθεσή μου. Και θυμίζω σε όλους μας και πάλι αυτό που πρόσφατα είπε ο Πιέρ Μοσκοβισή, ότι μπορεί εμείς να είμαστε η τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης. Είναι πολύ κρίσιμη η καιρή και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ σύντομη, ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε με την ησυχία μας αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Από το ΕΛΚ λοιπόν, ο κύριος Στορόγιαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι πως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε σε αυτή την ετήσια έκθεση για να δούμε τι γίνεται με τη φορολογική πολιτική των κρατών μελών. Προσωπικά θα ήθελα να υπογραμμίσουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το εξή. Το ότι είναι επίκαιρο το θέμα, το ότι είναι καυτό και ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τις πληροφορίες που θα φτάσουν από όλες τις πηγές. Τώρα, μιλώντας για τη φοροδιαφυγή, εκεί θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Και το τι θα γίνει με την επιθετική ε, φορολογική πολιτική που ακολουθούν ορισμένοι για να φορο, ε, για φοροαποφυγή. Τι απόκριση προσέφεραν τα κράτη-μέλη στις συστάσεις που απευθύνθηκαν σε αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έκαναν για τις τροποποιήσεις που τους προτάθηκαν ή τη φορολογική τους πολιτική, για παράδειγμα. Δηλαδή, μιλάω για τη μείωση του φορολογικού βάρους που αυτή τη στιγμή ε, επιβαρύνει την αγορά εργασία. Σε πολλά κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι φόροι ε, επί τη εργασίας είναι πραγματικά δυσβάσταχτοι. Άλλο ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, γιατί παρενθετικά θα πω ότι ελπίζω ότι αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών θα συμφωνήσουν για την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών για τα εισοδήματα και τα έσοδα των πολιτών μας στα άλλα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορούν ε, το θέμα της φοροαποφυγής να το καταπολεμήσουν καλύτερα, ε, πρέπει να σας πω πως ε, τελικά βλέπω δυστυχώς οι, οι διμερείς συμφωνίες να καθυστερούν πολύ. Για παράδειγμα, τι γίνεται με την Ελβετία. Μόνο δύο διμερείς συμφωνίες έχει υπογράψει μέχρι, μέχρι σήμερα για την διαφάνεια και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών πληροφοριών για τα εισοδήματα και τα έσοδα των Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι έχουν ανοίξει λογαριασμού στην Ελβετία. Δύο μόνο. Και αυτή ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία. Υπάρχουν χώρε όπω η Γαλλία, η Ισπανία κτλ. Ε, με τις οποίες τρέχουν διαπραγματεύσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι τρέχουν με το ρυθμό ε, του σαλγαριού. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό της φοροαποφυγής. Ε, κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να ζητηθούν ευθύνε. Οι πολίτες μας θα μας ρωτήσουν γιατί. Γιατί καθυστερούμε τόσο πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτούς, αυτά τα άτομα τα οποία ε, με επιθετικό τρόπο καταφέρουν να αποφύγουν τη φορολόγηση. Εκεί κάποια πρόοδος έχει ε, σημειωθεί γιατί και ο ΣΑ έχει λάβει κάποιες αποφάσεις σχετικές Θέλω να σας πω τι γίνεται στη χώρα μου για παράδειγμα. Εμείς έχουμε εταιρείε πολυεθνικές οι οποίες κάθε χρόνο ε, δηλώνουν ζημία και παρόλα αυτά φαίνεται ότι τα κέρδη μεγενθύνονται παράλληλα με αυτές τις ζημίες. Και παρόλα αυτά δεν χρεοκοπούν. Δεν δηλώνουν ε, ε, πως έπεσαν έξω. Γιατί αυτά τα οποία δηλώνουν στην πραγματικότητα δεν έχουν συμβεί. Αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει σε κάθε χώρα που έχουν οικονομικές δραστηριότητες να αναφέρουν ποια ήταν τα κέρδη τους στην συγκεκριμένη χώρα και παράλληλα με αυτό σε κάθε χώρα τι φόρο επί αυτών των κερδών κατέβαλαν. Θα πρέπει λοιπόν εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αμυνθούμε με στεναρότητα. Γιατί υπάρχει ένα θέμα υπέρ του οποίου έχουν στρατευτεί τα περισσότερα ε, αναπτυγμένα ε, κράτη. Δηλαδή, τον Ιανουάριο του 2015 οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν κέρδη και φόρους σε κάθε κράτος στις οποίες έχουν έδρα ή έχουν οικονομική δραστηριότητα. Εγώ θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια και με τους σκιώδες βεβαίως για να καταφέρουμε η έκθεση αυτή ε, να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αμποτέρχο από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομες παρατηρήσεις σε αυτή τη φάση. Αυτό που θα θέλαμε να γίνει στην εκθέση αυτή είναι να υπάρξει έμφαση στα εξή τρία σημαντικά ζητήματα για την φορολογία. Πρώτον, προτιμούμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονό ότι η φορολογία κατεξοχήν παραμένει μέρος της εθνικής αρμοδιότητας και πρέπει να παραμένει στα πλαίσια της εθνικής δικαιοδοσίας. Όμω, σε δεύτερη φάση, θα θέλαμε να υπάρχει συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και συντονισμό, καθώ υπάρχουν συγκεκριμένα ωφέλη που θα μπορούσαμε να αποσπάσουμε από την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη. Τρίτον, παρόλο που η προλογική πολιτική παραμένει εθνική αρμοδιότητα κατεξοχήν, είμαστε πρόθυμοι να ε, διασταυρώνουμε πληροφορίε ε, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να δώσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να τι ανταλλάσσουν. Αυτά σε αυτή τη φάση. Σας ευχαριστώ και ε, ευχαρίστω να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και τους σκιώδει εισηγητέ για την εξέβρεση λύσεων. Ευχαριστούμε τώρα για την άλλη κυρία Φαν Νόιερχόιζεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, νομίζω ότι και εγώ μπορώ να είμαι σύντομη. Για του φιλελεύθερου, η καταπολέμηση τη προδιαφυγή, τη φοροπάτη και των φορολογικών παραδείσων είναι ε, ύψιστη προτεραιότητα. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι οι εταιρείε και οι πολίτε ε, έχουν να αντιμετωπίσουν ίσου ε, κανόνε σε μια διεθνή αγορά και διαφανή βάση του διεθνού δικαίου. Δεν αρκεί να παραμένουμε στο γράμμα του νόμα, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται και το πνεύμα αυτού. Είναι προ όφελο των πολιτών και των κατών μελών να ανακόψουν την παράκαμψη του ε, φορολογικού συστήματος καθώς πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην ε, επιβολή, την ορθή επιβολή των ε, φόρων. Θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία των φορολογικών αρχών, ώστε οι μεγάλες πολυεθνικές να καταβάλουν το τίμημα που τους αναλογεί, όπως και οι περισσότεροι πολίτες. Θα θέλαμε επίση να μην υπάρξουν στρεβλώσει του ανταγωνισμού ε, που μπορεί να είναι επεζήμιες στι ευρωπαϊκέ εταιρείε και την ανάπτυξη με ένα κατάλληλο ε, ευεργετικό κλίμα. Η φορολογική πολιτική στα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι διαφανή και συνεκτική. Δεν ε, θέλουμε, δεν υπάρχει λόγος να καταπολεμήσουμε τον φορολογικό ανταγωνισμό, αλλά πρέπει να υπάρχουν χαμηλά επιτόκια με την μετατόπιση από την εργασία, τη φορολόγηση της εργασίας στην κατανάλωση. Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο τώρα είναι θέσεις εργασίας. Οπότε είναι ένα σημαντικό μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί. Και εγώ ευχαριστώ να συνεργαστώ ε, με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε. Και τώρα για την ΚΟΕ, ο κ. Βιέγκας. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την χειροπιαστή πραγματικότητα εντό τη οποία ζούμε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχουν φορολογικές ε, προσπάθειες ενοποίησης που τελικά βαρύνουν πάντα τους ίδιους, δηλαδή τους φορολογμένους. Είναι ο ευκολότερος στόχος. Είναι πιο εύκολο να επιβάλλεται φόρος επί του εισοδήματος ή ο φόρος προστιθέμενης αξίας στους πολίτες πρέπει να μην ξεχνάμε το σημείο αφετηρία στην αυτή η πραγματικότητα και ότι η λιτότητα έχει βαρύνει ακριβώ κυρίω του εργαζομένου. Αυτό ξεκινάει και από ένα πρότυπο, ένα μοντέλο που έχει επικρατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει ξεπεράσει κάθε άλλη προτεραιότητα, δηλαδή την απελευθέρωση των ε, κεφαλαίων και των συναλλαγών, των μετακινήσεών τους, κάτι που ουσιαστικά διευκολύνει αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαπάτη. Αυτό θα έπρεπε να είναι το σημείο αφετηρία του συλλογισμού μα. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν, αλλά τα ωραία λόγια δεν αρκούν. Ακούσαμε πολλά ωραία να λέγονται τις τελευταίες εβδομάδες και όχι μόνο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μεταφράσουμε αυτά τα λόγια και σε πράξεις. Διότι η απελευθέρωση της κυκλοφορίας των, κελαφέ, των, κεφαλαίων έχει γεννήσει ένα τέρας επί της ουσίας. Ένα τέρας που ας αναγκάζει σε κοινωνικό επίπεδο να αναζητούμε την αντιμετώπιση της φοροαπάτης ε, να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους φορολογικούς παραδείσους που δεν είναι κάτι το ε, άειλο και άπιαστο, είναι μέρη πραγματικά που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε την φοροαπάτη, τη φοροδιαφυγή, τις τραπεζικές αγορές και μεταξύ πολλών άλλων θα έπρεπε να εφαρμόζουμε το, τις αρχές, την αρχή του οικολογικού φόρου όπως ο φόρος το BIN να επιβληθεί ένας φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Κάτι που δεν θα διορθώσει, δεν θα είναι μια μαγική λύση στην αρνητική πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον θα προβλέψει μια κάποια φορολογική δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις. Ευχαριστούμε για τους, green, για τους πράσινους, η κυρία Σκάτ. Ε, νομίζω το πιο σημαντικό που ακούσαμε και το πιο θετικό ήταν αυτό που είπε ο κ. Μοσκοβίτση την περασμένη, την περασμένη εβδομάδα στην πρόασή του. Ότι χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση στι φορολογική πολιτικέ και ότι θέλει στενότερη συνεργασία μαζί μα για να πετύχουμε αυτόν τον κοινό στόχο. Νομίζω ότι όλοι εδώ στην Επιτροπή συμφωνούμε ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα και θα θέλαμε να κάνουμε κάποια θετικά βήματα προ αυτή την κατεύθυνση τα επόμενα χρόνια. Επιτέλου, οι πράξει να συνοδεύσουν τα λόγια μα. Για του πρασίνου, ο φόρο είναι το τίμημα που πληρώνουμε για να ζούμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Είναι λοιπόν μάλλον καθόλου αξιέπαινο το να αποφεύγει κανείς να πληρώνει τους φόρους του. Ε, η στήριξη του κυρίου Μοσκοβησί για, την, για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ήταν κάτι που πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό, διότι τα κονδύλια που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από ένα τέτοιο φόρο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ένδυας και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Αυτό είναι λοιπόν κάτι στο οποίο και εμείς μπορούμε να προσχωρήσουμε. Επίσης, στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις ματοχές και τα τραπεζικά παράγωγα, τα σχετικά προϊόντα στην φορολόγηση. Να μην πληγεί η σταθερότητα της, ε, της σχετικής αγοράς βέβαια, αλλά τουλάχιστον να αντλήσουμε κάποιες πηγές ε, που κονδυλίων που αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. Βεβαίω, θα θέλαμε και άλλε χώρε να στηρίξουν το φόρο χρηματοδοτικών συναλλαγών, καθώ υπάρχουν πολλέ, όπω και δική μου, που ακόμη δεν δέχονται αυτή την επιλογή. Ε, βλέπουμε πάντω να υπάρχει σχετική συμφωνία στα τρία αυτά σημεία και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε και την άγρα χαμηλών φορολογικών επιτοκίων με τη μεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μια σταθερότητα και μια ενοποίηση για να μπορέσουν και οι πολίτες να ε, προστατευτούν. Και επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε και τους σχετικούς κανόνες της Γενικής Διεύθυνσης ε, Φόρων ε, με παρόμοιες, με σχετικές έρευνες που βλέπουμε να διεξάγονται αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο ή τις κάτω Πρέπει να έχουμε ασφαλή φορολογικά στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη και να συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές. Δεν θα πρέπει απλώς να έχουμε κατά νου ένα παιχνίδι θόνου μεταξύ μας που τελικά δεν ωφελεί κανέναν. θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους φόρους των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ε, για τους ε, προσωπικούς φόρους θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ανταλλαγής, αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, όπως προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οδηγία της για τη διοικητική συνεργασία. Νομίζουμε πληροφορίες κατόπιν αιτήματος η κατακράτηση στοιχείων όπως κάνουν αυτή τη στιγμή η φορολογική παράδειση όπως το Λουξεμβούργο δεν είναι κάτι που μπορεί, θα πρέπει να διατηρηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε εδώ αποτελεσματικά με τους υπόλοιπους σκιώδεις ώστε να αναπτύξουμε ένα φορολογικό σύστημα που να ωφελεί τους πολίτες και να επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ευχαριστώ. Από την EFTD δεν υπάρχει ομιλητή, οπότε θα δώσω ξανά το λόγο στην εισηγήτρια για να κλείσουμε. Well, I think, uh, Thank Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι είναι κοινέ οι απόψεις, υπάρχει συναντήληψη. Ε, θα ε, συνεργαστούμε για τα θέματα αυτά τους επόμενους μήνες και ελπίζουμε με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι μέχρι σήμερα. Είναι κρίσιμη η καιρή και η στιγμή και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Οι πάντες περιμένουν την έκθεση αυτή και θα πρέπει να αρχίσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η νέα πολιτική. Σας ευχαριστώ και θα το ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Ε, ο Πρόεδρος, εδώ τελείωσε ο χρόνος μας. Κύριε Μαριά, μας ζήτησα το λόγο την ώρα που μιλούσε η κυρία Καηλή. Ναι, αλλά γνωρίζετε ε, τους κανόνες. Κάτσε έχουμε και δίνουμε όταν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς ε, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας στην ψηφοφορία. Α, κατάλαβα. Πληρώνουμε το τίμημα της δημοκρατίας με χρόνο. Ε, ωραία. Ε, εδώ η συνεδρίασή μας. Λύεται η συνεδρίαση. Επόμενη συνεδρίαση προπαρασκευαστική για τα μέλη της ΕΚΟΝ για την ε, Κεντρική Τράπεζα και τα τεστ ατοχής στην ίδια αίθουσα εδώ. Θα έχουμε εξωτερικούς ομιλητές, ε, εκλεκτούς που τους έχουμε προσκαλέσει να συμμετάσχουν. Σε λίγα λεπτά.